Ladies and gentlemen, after... Κυρίες και κύριοι, μετά από αυτό το θαυμάσιο βίντεο, έχω την τιμή και την ευχαρίστηση να σας καλωσορίσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από πλευρά του Προέδρου Αντώνιο Ταγιάννη, που θα μας κάνει μια κεντρική ομίλη αργότερα. Χαίρομαι πολύ που ανοίγω αυτή τη ε, συνδιάσκεψη για τους ωκεανούς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πρόσκληση του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής. Μπορώ να σας πω ότι θα μεταφραστεί σε 23 γλώσσες. Οπότε αν θέλετε να ακούσετε οποιαδήποτε διερμηνία μπορείτε να το κάνετε και επίσης πρέπει να σας πω ότι όπως πολύ συχνά στο Κοινοβούλιο εκπροσωπούνται και τα δύο φύλλα εξίσου. Η διάσκεψη διοργανώνεται από τον πρόεδρο Ταγιάννη με τις αρμόδιες επιτροπές την Επιτροπή Περιβάλλοντος, την Επιτροπή αλληλεία και την Επιτροπή Έρευνας και Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ιδιαίτερα με τη Γενική Διεύθυνση για τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και άλλες υπηρεσίες Κομισιόν. Και καλωσορίζω και τους επιτρόπους Βέλα και Μοέντας που ε, συμμετέχουν στη διοργάνωση και σε αυτήν την ανακτήρια συνεδρίαση. Παράλληλα, είναι θαυμάσιο που είναι εδώ και εκπρόσωποι της νέας γενιάς, α, και από την άλλη πλευρά έχουμε δύο εκπροσώπους ε, νέων και πολλούς άλλους ε, στην αίθουσα. Γι' αυτό καλωσορίζω θερμά τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό από τα ευρωπαϊκά σχολεία της Βρυξέλλης. Μπορείτε να σηκώσετε τα χέρια σας. Ευχαριστώ. Καλώς ορίζουμε τη νέα γενιά. Αυτό καταδεικνύει ότι εκεί ανήκει το κλίμα, είναι στο κέντρο της προσοχής της νέας γενιάς και αυτό είναι θαυμάσιο. Κυρίες και κύριοι, η θαλάσσια πολιτική έχει διάφορες πλευρές. Δεν είναι δυνατόν να τα συζητήσουμε όλα σε μία μόνο εκδήλωση μισή μέρα, Αλλά κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Και οι ομιλητές προέρχονται από διαφορετικά επαγγελματικά πεδία και ασχολούνται με διάφορες πλευρές της αλλαγής πολιτικής, έρευνα, οικονομικά θέματα και συμμετοχή των πολιτών. Και έχουμε τρεις συζητήσεις στο τραπέζι. Πρώτον, η διακυβέρνηση των ωκεανών για το μέλλον. Ε, τώρα δεν θα μιλήσω για συγκεκριμένου ομιλητές αλλά θέλω να καλωσορίσω θερμά την πρώην Επίτροπο για την Αλληλεία και τις θαλάσσιες υποθέσει Μαρία Δαμανάκη. Νομίζω ότι σε είδα να κάθεσαι εκεί, σε καλωσορίζουμε. Η κυρία Δαμανάκη ήταν υπεύθυνη για τη μεταρρύθμιση της κοινή αλληλευτικής πολιτική που ήταν ένα μεγάλο βήμα προόδου για την Ευρώπη. Η δεύτερη συζήτηση θα ασχοληθεί με τι προκλήσει για να υπάρξουν υγιεινείς και καθαρές, ε, συγγνώμη, ε, υγιείς και καθαρές θάλασσες για να αντιμετωπίσουμε τη μόλυνση. Και θα συζητήσουμε την μελλοντική πορεία στο τρίτο γύρο μιλητών για να προωθηθεί η γαλάζια οικονομία όχι μόνο στους παραδοσιακούς τομείς αλλά και αναδυόμενους νέους τομείς όπως η παραγωγή φυκιών και η παραγωγή ενέργειας από τις θάλασσες. Ε, σε κάθε συζήτηση θα έχουμε ε, την Προεδρία του Προέδρου ή Αντιπροέδρου των Αρμοδίων Επιτροπών και άλλοι ευρωβουλευτές θα κάνουν και σύντομες δηλώσεις. Αγαπητοί φίλοι, δεν έχουμε χρόνο για να κάνουμε διάλειμμα, αλλά αν κατόπιν ε, βρείτε χρόνο, μπορείτε να δείτε τις εκθέσεις που έχουμε και μπροστά και στις δύο πλευρές του ημικυκλίου. Θα δείτε καταπληκτικά παραδείγματα προγραμμάτων που χρηματοδότησε η Ένωση όπως ο Κοπέρνικος, που ασχολείται ιδιαίτερα και με θαλάσσιες υποθέσεις, ή το πρόγραμμα Μαρίνα και η υπεύθυνη κατάρτιση για τη γνώση των ωκεανών. Και Σήμερα συμμετείχα σε ένα διάλογο για τους ωκεανούς όπου συζητήσαμε με νέους επαγγελματίε του τομέα το Marina και το Responsible και το μήνυμά τους είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε στις καθημερινές συζητήσεις ε, των συμπολιτών μας να αναφέρω τα θέματα των ωκεανών. Ακόμη δεν το έχουμε καταφέρει. Αυτό το, συζητάμε τουλάχιστον όλα μέλα. Τα τελευταία δύο χρόνια επιτύχαμε να συζητηθούν πολύ περισσότερο οι ωκεανοί και οι θάλασσες και να γίνουν προτεραιότητα. Όχι μόνο λόγω της μόλις από τα πλαστικά, δυστυχώς αλλά ευτυχώς και για άλλους λόγους. Είχαμε μεγάλες διασκέψεις όπως ο ωκεανός μας, τον Παλί, φέτος ε, στην Νορβηγία και επίσης μικρές πρωτοβουλίες που οργανώνουν διάφορες μη κυβερνικές οργανώσεις για τον καθαρισμό στις παραλίες. Ε, έχουν γίνει λοιπόν οι θάλασσες θέμα παντού. Δεν το γνωρίζουν ακόμη όλοι, αλλά έχουμε κάνει πολλά. Καλό λοιπόν θα ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δημιουργήσει μια επιτροπή για τις θαλάσσιες υποθέσεις. Μάρε, όπου να μπορούμε να συζητήσουμε όλα τα θαλάσσια θέματα. Και οι διασκέψεις που κάνουμε τώρα βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα άλλο καλό παράδειγμα θα ήταν το... η διαπολιτική ομάδα που έχουμε για τις θάλασσες, τους ωκεανούς και τα νησιά και τις παράκτη περιοχές. Το ακρονίμιο είναι ΣΥΡΙΚΑ. Το δημιουργήσαμε το 2014 για νέα πλατφόρμα για τα θαλάσσια θέματα και για να εμπλακεί σε αυτή τη συζήτηση συνολικά η κοινωνία μας, οι οργανώσεις, η κοινωνία των πολιτών κτλ. Γιατί η ωκεανή και η θαλάσσια πολιτική είναι τόσο σημαντική για μας. Γιατί ζούμε σε έναν γαλάζιο πλανήτη. 70% της επιφάνειας του πλανήτη μας είναι νερό και είναι ζωτική για το κλίμα. Διότι δεσμεύουν το διοξείδιο του άνθρακα και παράγουν οξυγόνο. Κάθε δεύτερη αναπνοή μα περιλαμβάνει οξυγόνο που έχει παραχθεί στου ωκεανού και είναι πολύ σημαντική για το μέλλον τη ανθρωπότητα. Αυξάνεται ο πληθυσμό μα και χρειάζονται τροφή και από τους ωκεανούς, ενέργεια, μπλε, βιοτεχνολογία και βεβαίως ε, οι θαλάσσιες μεταφορές είναι το 90% των ε, μεταφορών, αλλά απειλούνται οι ωκεανοί. Χρειαζόμαστε υγιείς ωκεανούς για το μέλλον της ανθρωπότητας. Αυτό είναι σημαντικό φυσικά και για μας τους Ευρωπαίους. Η Ευρώπη είναι θαλάσσια ήπειρος. Η ακτογραμμή μας είναι 7 ε, φορές μεγαλύτερη από την ακτογραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών και μόνο πέντε κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν ακτογραμμή και είμαστε ηγέτες στην ε, πράσινη αυσιπλοεία, την ενέργεια από τα κύματα, από τα παλαιριακά κύματα και από τις ε, υπεράκτιες ε, ανεμογεννήτριες. Έχουμε εδώ τον καθηγητή Χέρτσιγκ που θα μας μιλήσει αργότερα για τα θέματα αυτά. Αλλά δεν χρειαζόμαστε μόνο περισσότερη έρευνα. Ξέρετε, ξέρουμε περισσότερα για τη σελήνη από ό,τι για τα βάθη των ωκεανών. Θέλουμε πολύ περισσότερα στοιχεία για τους ωκεανούς. Θέλουμε να υπάρχει ανταλλαγή των ε, αποτελεσμάτων της έρευνας. Και πρέπει η επιστήμη να είναι σε σωστή επαφή με το λαό. Πρέπει να γνωρίζει ο λαός, οι συμπολίτε μας, τα των ωκεανών. Γι' αυτό πιέζουμε για πιλωτικά προγράμματα, για την γνώση για τις θάλασσες και μόνο πριν από μερικές χρόνιες έγινε μια έκκληση από τη Γενική Διεύθυνση ΜΑΡΕ για τα θαλάσσια θέματα. Και κάτι πολύ σημαντικό. Και η UNESCO προετοιμάζει τη δεκαετία για την ε, επιστήμη των ωκεανών που θα ξεκινήσει το 2021. Θα μα πει ο κ. Διαμήνιν περισσότερα γι' αυτά. Αγαπητοί φίλοι, η πολιτική των θαλασσών μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μακρά παράδοση. Το Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συζήτησαν την ολοκληρωμένη ε, θαλάσσια πολιτική, την μπλε οικονομία, την κοινή γεωρική πολιτική, την ε, διακυβέρνηση των ωκεανών. Βγάλαμε πρόσφατα ένα φυλάδιο και πρόσφατα είχαμε και οδηγίες για τα πλαστικά ούτως ώστε να καθαρίσουμε τους ωκεανούς μας. Όλα αυτά τα κάναμε σε στενή συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμών της Ένωσης. Το Συμβούλιο επίσης, λοιπόν, μαζί με το Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πολλά για να προωθηθούν τα θέματα αυτά, αλλά πάντα στηρίχθηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και τώρα Τώρα πρέπει να εφαρμόσουμε στα κρατη αυτά που αποφασίστηκαν. Είναι ένα ακούγεται εύκολο, αλλά δεν είναι πάντα εύκολο. Και επίση οι νέοι πρέπει να είναι διατεθειμένοι να επιλέξουν μπλε σταδιοδρομίε για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Σε στενή συνεργασία με οργανισμούς όπως ο ε, οργανισμό που θέλει να σταματήσουν οι πλαστικέ σακούλες και διάφορε άλλε πρωτοβουλίε. Ε, που κάνουν πορείες για το περιβάλλον ή με νέους καινοτόμους ηγέτες που ασχολείται με την αντιμετώπιση των σκουπιδιών στον ειρηνικό. Η Ένωση είναι παγκόσμια πρωτοπορία στην έρευνα και καινοτομία. Πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτά τα προτερήματά μας για να επιτύχουμε μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία. Και χρειαζόμαστε οπωσδήποτε στο επόμενο πλαίσιο ε, για την έρευνα να έχουμε ειδικό κεφάλαιο για τις θάλασσες και τους ωκεανούς. Επίκυνται οι ευρωεκλογέ, το ξέρετε. Έχουμε λοιπόν αυτή την εκδήλωση για το μέλλον του γαλάζιου πλανήτη. Οι ωκεανοί βέβαια δεν ε, ψηφίζουν, ε, δεν είναι ψηφοφόροι, αλλά είναι πολύ σημαντικοί για μας. Κάποιο που τα ξέρει όλα αυτά, τη σημασία των ωκεανών λοιπόν, θα συμφωνήσει απόλυτα νομίζω ο οποίο φιλοξένησε την διάσκεψή μα για του ωκεανού στη Μάλτα το 2017 είναι ο Επίτροπός μας για θέματα άλλης Καρμίνου Βέλα, στον οποίο θα δώσω τώρα το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι Γεζίνε, Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ Επίτροπε Κάρλος, αγαπητή Τέος Επίτροπε Μαρία, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί προσκεκλημένοι, πρώτα απ' όλα θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήρθατε εδώ να συζητήσουμε μαζί το μέλλον του γαλάζιου πλανήτη μας. Όπως πολλοί Ευρωπαίοι, μεγάλωσα και εγώ δίπλα στη θάλασσα κυριολεκτικά και έχω πάρα πολύ ε, θερμές αναμνήσεις από την παιδική μου ηλικία και τα καλοκαίρια που περνούσα στις παραλίες, ε, παρθένα νερά, πολύ ωραίες αναμνήσεις ε, και όσο μεγαλώνω τόσο τις θεωρώ πιο σημαντικές αυτές τις αναμνήσεις. Είδα όμως και αρνητικά να συμβαίνουν πίεση στα οικοσυστήματα και στους διάφορους πόρους. Έχω ακούσει φίλους μου ψαράδες να παραπονούνται ότι δεν έχουν τόσα ψάρια να ψαρέψουν. Είδα επίσης ε, να γίνεται λόγος για την αλλαγή του κλίματος, την υπεραλίευση, την ρήπανση. Ε, μπαίνουν στο προσκήνιο αυτές οι συζητήσεις και όλα όσα συμβαίνουν σήμερα μας κάνουν να αντιληφθούμε ότι πράσινο και γαλάζιο πρέπει να συμβαδίζουν. Από τότε που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, πριν πέντε χρόνια περίπου, εργάστηκα σκληρά για να περάσω αυτό το μήνυμα και για να δημιουργήσω ένα συνασπισμό για υγιείς παραγωγικές θάλασσες και ωκεανούς. Είτε εδώ, ε, στη χώρα μου, είτε στο εξωτερικό. Συμμαχία από ακτιβιστές, πολιτικούς, επιστήμονες, ε, πολίτες, νέους ανθρώπους που τους ενδιαφέρει το μέλλον που θα κληρονομήσουν μια μέρα από εμάς αυτό το γαλάζιο πλανήτη. Χαίρομαι πολύ λοιπόν που βλέπω να είναι γεμάτη σήμερα η αίθουσα γιατί αυτό δείχνει ότι υπάρχει όλο και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τη σημασία των ωκεανών, για την οικονομία, για το κλίμα μας, αλλά πάνω απ' όλα για την επιβίωσή μας πολύ απλά. Και είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος για τα επιτεύγματα της Ένωσης τα τελευταία πέντε χρόνια. Πρώτα απ' όλα Έχουμε κανόνες που περιορίζουν τη χρήση των πλαστικών μιας χρήσης. Έχουμε στόχους ανακύκλωση δεσμευτικούς. Όλα αυτά καθιστούν την Ένωση παγκόσμιο πρωταγωνιστή για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων. Δεύτερον, έχουμε ορίσει πάνω από το 10% ε, των θαλάσσιων περιοχών, των ακτογραμμών, ω προστατευόμενε θαλάσσιε περιοχέ, δύο χρόνια πριν από την λήξη τη Διεθνού Προθεσμία του 2020. Και αυτό συνεισφέρει στο να έχουμε καλή κατάσταση περιβαλλοντική για τους ωκεανούς μας σύμφωνα και με το ενιαίο ε, θαλάσσιο πλαίσιο, τη σχετική οδηγία. Τρίτον, πιέζουμε για πιο βιώσιμη αλληλεία και αυτό αποδίδει σε πολλές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, η αλία είναι σε πολύ καλή κατάσταση, στην καλύτερη εδώ και δεκαετίε. Τα αλλιεύματα, ε, τα οποία αλλιεύονται σε βιώσιμα επίπεδα, έχουν διπλασιαστεί. 51 ήδη φέτο σε σχέση με 27 όταν αναλάβαμε καθήκοντα και 5 μόλι πριν από 10 χρόνια. Τέταρτον, αναδυόμενοι τομεί ε, τη ε, βιώσιμη θαλάσσια οικονομία είναι πλέον στο προκείμενο. Η ενέργεια από του είναι ένα καλό παράδειγμα. Και έχει λάβει και σημαντική χρηματοδότηση για έρευνα, για πειραματισμό. Είναι ένα τομέα τραχαίως αναπτυσσόμενο και περνάμε στην φάση πρώτη ε, διάθεση στο εμπόριο. Επίση, υπάρχουν και άλλες καινοτόμε θαλάσσιε επιχειρήσει ε, και κλάδοι που θα ε, βοηθηθούν από την πλατφόρμα που θα δρομολογήσουμε αργότερα φέτο. Επίση, τα δύο τελευταία χρόνια επενδύσαμε πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ στην έρευνα, τη θαλάσσια έρευνα συγκεκριμένα, παραδείγματι το μικρό του τους ενδεχόμενους κινδύνους ε, των μικροπλαστικών για τη θαλάσσια ζωή αλλά και για την ανθρώπινη υγεία. Και γνωρίζω πως ο συνάδελφός μου Κάρλος Μοέδας θα πει περισσότερα για το θέμα αυτό σε λίγο. Δεν έχουμε όμως ε, περιορίσει τις φιλοδοξίες μας μόνο στην Ευρώπη γιατί η ε, ωκεανή είναι μια κοινή ευθύνη παγκόσμια. Χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να αναγγείλω ότι μόλις δημοσιεύσαμε την πρώτη έκθεση πρόοδου για το τι έχει πράξει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιώσει τη διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία καταγράφει το τι πετύχαμε από τότε που εγκρίναμε το θεματολόγιο για μια καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη διακυβέρνηση των ωκεανών τον Νοέμβριο του 2016. Πρόκειται για ένα θεματολόγιο με 50 δράσει ε, που έχει αναζωογονήσει τη διεθνή συνεργασία. Είναι ένα θεματολόγιο που σφυριλατεί και παγιώνει την φήμη τη Ευρωπαϊκή Ένωση ενό ε, ως ένα εταίρο αξιόπιστο. Παρέχουμε τεχνική βοήθεια, χρηματοδότηση για βιώσιμη δράση και οικονομική ανάπτυξη και είμαστε στην κορυφή. 600 εκατομμύρια ευρώ περίπου έχουμε ε, διαθέσει για τη στήριξη της αλίας και της ηχθειοκαλλιέργειας, για την υποστήριξη των περιοχών που βασίζονται στην αλία, για πιο καθαρές θαλάσσιες μεταφορές και για βελτίωση των λιμενικών υποδομών και της θαλάσσιας ασφάλειας στις χώρες εταίρους. Βοηθήσαμε σημαντικές αλληλευτικές δυνάμεις να βελτιώσουν τα συστήματα ελέγχου ώστε να μπορεί να καταπολεμηθεί καλύτερα η παράνομη αλία και πιο αποτελεσματικά ε, με το σύστημα της χίτρινης και της ε, κόκκινης κάρτας. Επίσης έχουμε διμερείς εταιρικέ σχέσεις ε, με φορείς σημαντικούς χώρες όπως η Κίνα, ο Καναδάς. Επίσης έχουμε ολοκληρώσει μια νέα λευτική συμφωνία με την Αρκτική για να μην υπάρχει ανεξέλεγκτη εμπορική αλληλεία στον Αρκτικό ωκεανό στα Επίσης ε, προωθούμε βιώσιμες ε, γαλάζιες οικονομίες και εντό ε, τη Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε άλλες τρίτες χώρες νησιωτικέ μέσω των αρχών της θαλάσσιας βιώσιμης οικονομίας για να προωθήσουμε βιώσιμη οικονομία στο ωκεανούς. Επίκυνται ευρωεκλογέ. Είμαι πεπισμένος περισσότερο από ποτέ ότι οφείλουμε να πούμε στους πολίτες τι κάνει για αυτού η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι κάνει για τις τοπικέ κοινότητε, για τι οικογένειε, για το μέλλον τους. Και ο ωκεανό είναι το καλύτερο μέρο να ξεκινήσει κανεί. Όπω ε, ε, αρέσει και τα λέει άλλωστε και ο πρόεδρο Γιούγκερ, θέλουμε να είμαστε μεγάλοι στα μικρά πράγματα. Και τι πιο μεγάλο υπάρχει από τον ωκεανό. Ε, περάσει λοιπόν αυτό το μήνυμα προς τα έξω για να μάθει ο κόσμος ε, πώς εργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τις ε, θαλάσσιες περιοχές ε, για ένα γαλάζιο πλανήτη, τον δικό μας γαλάζιο πλανήτη για το μέλλον μας, το δικό μας μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ Καρμένου. Στη συνέχεια μπορώ να δώσω το λόγο στο Συμβούλιο. Ξέρετε ότι έχουμε τρία θεσμικά όργανα, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τώρα η Ρουμανία έχει την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Αντριάννα Πέτκου είναι αναπληρώτρια υπουργό Υδάτων και Δασών. Νομίζω περισσότεροι χρειαζόσαστε ακουστικά διότι η προσκεκλημένη μας θα μιλήσει στα ρουμανικά. Έχετε το λόγο. Thank you, Ευχαριστώ, Γεζίνε. Κύριοι Επίτροποι, κύρια Πρόεδρε, αγαπητά μέλη, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διοργάνωση αυτής της εξαίρετης διάσκεψης μέσα στα πλαίσια των προσπαθειών μας να σώσουμε τους ωκεανούς και τις ανοιχτές θάλασσες έτσι ώστε να υπάρχει βιώσιμη ανάπτυξη και δραστηριότητες από τις ε, οποίες εξαρτώμεθα. Θεωρούμε ότι οι ωκεανοί και οι ανοιχτές θάλασσες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του παγκόσμιου οικοσυστήματος. Οι ωκεανοί μας δίνουν χώρο, πόρους, ενέργεια και τροφή για την ανθρωπότητα. Γι' αυτό οι ωκεανοί και οι θάλασσες μπορούν να εξαλείψουν τη φτώχεια προσφέροντας νέες θέσεις βιώσιμης εργασίας. Αυτό όμως το βασικό στοιχείο ρύθμισης σημαίνει ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον και να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της βιωσιμότητας για τους ωκεανούς. Αυτό αποτελεί υποχρέωσή μας, έτσι ώστε να μην ακολουθήσουν φθήνουσα πορεία οι ωκεανοί καθώς και το θαλάσσιο περιβάλλον που είναι κλειδί για τις πολιτικές μας. Εμείς προσδίδουμε μεγάλη, σημασία στην προστασία των θαλασσών. Για μας η Μαύρη Θάλασσα προσδίδει πόρους και αποτελεί ένα εξαίρετο οικοσύστημα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι ανθρωπογενείς πιέσεις από 200 δις ανθρώπους ως προς την παράνομη δράση τους, καθώς και τη μόλυνση της θάλασσας. Θα πρέπει να προωθήσουμε την βιώσιμη αλληλεία και να διασώσουμε το θαλάσσιο οικοσύστημα μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης των παρακτήων περιοχών, παρά τις εθνικές μας προσπάθειες, η προστασία των θαλασσών δεν μπορεί να γίνει χωρίς την περιφερειακή προσέγγιση που βασίζεται στη σύμβαση για την προστασία της μαύρης θάλασσας κατά της μόλυνσης. Γι' αυτό θα θέλαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει εταίρος και αναπόσπαστο μέρος αυτής της σύμβασης. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η θα πολλές πιέσεις ως προς την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Τα πλαστικά και τα μικροπλαστικά αποτελούν μόνιμη απειλή του θαλάσσιου περιβάλλοντος γιατί δεν υπάρχει σωστή διαχείριση θαλάσσιων αποβλήτων. Το θέμα των θαλασσίων αποβλήτων είναι περίπλοκο λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα καθώς και των ιδιοχαρακτηριστικών των θαλάσσιων περιοχών. Η επίλυση αυτών των θεμάτων σημαίνει προσπάθειες σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Γι' αυτό οι περιφερειακές συμβάσεις έχουν μεγάλη σημασία για την εφαρμογή των θαλάσσιων στρατηγικών στους ανοικτούς ωκεανούς. Η σύμβαση που αφορά τη Μαύρη Θάλασσα αναφέρεται στην ε, καταπολέμηση των θαλασσίων αποβλήτων και οι όμορες περιοχές καταβάλουν επίσης πολλές προσπάθειες. Η αύξηση των ε, πλαστικών θα πρέπει να καταπολεμηθεί, να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τα συλλέξουμε μέσα στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας. Έχει μεγάλη σημασία η αποθήκευση, διακίνηση και η ανακύκλωσή τους. Γι' αυτό δεν θα πρέπει να αποτεφρώνονται αλλά να ανακυκλώνονται τα πλαστικά. Θα πρέπει η ανακύκλωση να είναι σημείο κλειδί για την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος. Να επικεντρωθούμε στη γενική πρόληψη ως προς τα απόβλητα και τη σωστή διαχείρισή τους. Γι' αυτό προβάλλουμε και εταιρικέ σχέσεις. Όμως ε, θα πρέπει να έχουμε υπόψη και την κατανάλωση σε εθνικό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τη μόλυνση από τα πλαστικά και μικροπλαστικά, αυτό το θέμα θα απασχολήσει και το άτυπο συμβούλιο στις 20 και 21 Μαΐου στο Βουκουρέστι. Επίσης, σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να προγραμματίζουμε και να διαχειριζόμαστε τις οικονομικές δραστηριότητες στις παράκτιες περιοχές και να ανταλλάσσουμε πληροφορίες καθώς και να έχουμε συμμετοχή του κοινού. Να λάβουμε υπόψη τις κλιματικές αλλαγές που οδηγούν στην θέρμανση των ωκεανών και έχουν επίπτωση στις παράκτιες περιοχές. Η Ρουμανία έχει προβάλει ένα master plan για την προστασία των παρακτίων περιοχών της Μαύρης Θάλασσας, έτσι ώστε να σταματήσει και η διάβρωση των ακτών. Και αυτό αφορά και τη βιωσιμότητα των οικισμών κοντά στη θάλασσα. Επίσης, το Δέλτα του Δούναβη μας έχει απασχολήσει μέσα στα πλαίσια της διαχείρισης αυτής της ε, μεγάλης ε, λεκάνης απορροής και αυτό αφορά και τα παράκτια ε, ύδατα. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα θρεπτικά στοιχεία διατροφής που υπάρχουν στον Δούναβη και στην λεκάνη του Δούναβη που μειώνονται λόγω του ευτροφισμού. Θα πρέπει να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες για το οικοσύστημα αυτό της Μαύρης Θάλασσας με βάση την οδηγία πλαίσιο της στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θαλάσσιο περιβάλλον. Υπάρχει μία ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείριση των ωκεανών. Αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί για την βιωσιμότητα των οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών για να λάβουμε υπόψη τις κλιματικές αλλαγές και την προστασία της βιοπικιλότητας. Είμαι πεπισμένη ότι αυτή η διάσκεψη θα επιτρέψει να επιτελεστεί πρόοδος μέσα στα πλαίσια της βιώσιμης χρήσης ωκεανών και θαλασσών. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτός ο ρουμανικός οδικός χάρτης είναι πολλά υποσχόμενος σε συγχαίρω. Αν κάνετε όλα αυτά που έχετε προγραμματίσει, θα βοηθήσετε πολύ στην υγεία των ωκεανών. Επόμενος ομιλητής, ο Επίτροπος Κάλλος Μουέντας, που είναι αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία. Και, ε, όπως ξέρετε, ήδη έχουμε πει ότι 500 εκατομμύρια θα πάνε σε ειδικά προγράμματα έρευνας. Αλλά θα συμφωνείτε, κύριε Πίτροπο, ότι θα έπρεπε να είναι και περισσότερα, έτσι δεν είναι, θα ήταν καλύτερα. Έχετε τον λόγο παρόλα αυτά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και πρώην συνάδελφοι Καρμένου και Μαρία, και κάθομαι εκεί που ε, ήσασταν κι εσείς. Κάθε μέρα, δηλαδή το γραφείο μου είναι εκεί που ήσασταν εσείς, οπότε καταλαβαίνω και το δικό σας το καθήκον. Κοίταζα το κοινό και βλέπω τόσους νέους Νομίζω ότι η δική σας η γενιά, η νεότερη γενιά, είναι τόσο τυχερή. Είστε η γενιά που θα δει η επιστήμη να κάνει καταπληκτικά πράγματα, όπως και η τεχνολογία. Θα δείτε θεραπείες ε, για ασθένειες που ακόμη σήμερα δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε. Θα δείτε η κβαντική υπολογιστική να αλλάζει τον τρόπο λειτουργία των υπολογιστών. Αλλά θα αντιμετωπίσετε και μεγάλες προκλήσεις. Και η πρόκληση που συζητάμε σήμερα εδώ είναι μία από τις κυριότερες που έχετε ενώπιόν σας. Οπότε απευθύνομαι σε εσά για να σας πω ότι μετά από πέντε χρόνια εργασίας ως Επίτροπος και ταξιδεύοντας στην Ευρώπη, συναντώντας υπουργούς, πρωθυπουργούς, ε, σημαντικές προσωπικότητες. Όμως, ε, όταν σκέφτομαι την πενταετία που πέρασα, κυρίως θυμάμαι τους νέους που συνάντησα. Και ένα από τα άτομα που με ενέπνευσαν είναι ένας ε, ιδιαίτερα νέος. Ένας νέος που λέγεται Boyan Slad. Ο Boyan Slad είναι Ολλανδός. Όταν ήταν 16, φανταστείτε το, μόλις 16, πήγε στην παραλία στην ε, Μεσόγειο και είδε πολλά πλαστικά σκουπίδια και είπε «Μα τι έσχος είναι αυτό, κάτι πρέπει να κάνω». Και αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της γενιάς σας και της δικής μου. Η γενιά σας κάνει πράγματα. Καταλαβαίνει ότι ο ρόλος της δεν είναι απλώς να βρει μια δουλειά, να πάει στο πανεπιστήμιο και τέτοια. Είναι να αλλάξει τα πράγματα. Και η ιστορία του Boyan Slug, η ιστορία της γενιάς σας, είναι ότι ένας νέος, 16 ετών, να θεωρεί ότι είναι δουλειά του να καθαρίσει τις παραλίες και τους ωκεανούς. Και ε, ορισμένοι του λένε, κοιτάξτε, ε, υπάρχουν τόσες τεχνολογίες που μπορούν να μας βοηθήσουν να καθαρίσουμε τους ωκεανούς. Και ο Μπόιαν λέει, μα αυτοί απλώς ανακυκλώνουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να μην μπαίνουν ε, τα πλαστικά στον ωκεανό. Και εφήβρε μια νέα τεχνολογία που χρησιμοποιεί τα ρεύματα στη θάλασσα για να γίνει κάτι που πολλοί μηχανικοί και πολλοί άλλοι ειδικοί το συζητούσαν αλλά εξέταζαν τα θέματα με συμβατική άποψη. Ο Μπόγιαν προτείνει μια εντελώ διαφορετική προσέγγιση. Και αν επιτύχει σε αυτό που επιδιώκει, και βεβαίω ορισμένοι αμφιβάλλουν αν θα επιτύχει, αν είναι σωστή αυτή η τεχνολογία. Αλλά δύο πράγματα που έκανε είναι θεωρώ πολύ σημαντικά. Πρώτον, θεωρεί ότι είναι καθήκον του να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, αποστολή του. Αναλαμβάνοντας αυτή την αποστολή, κατάφερε να ε, βάλει τη συζήτηση αυτή στο επίκεντρο της προσοχής της κοινή γνώμης. Πριν από 15 χρόνια, αν σκεφτούμε πώς ήταν η συζήτηση, θα καταλάβετε ότι η κατάσταση έχει αλλάξει πολύ. Αλλά παρόλα αυτά, ε, μπορεί να έχει αλλάξει η κατάσταση στην κοινή γνώμη, αλλά η κατάσταση των ωκεανών δεν έχει αλλάξει. 8 εκατομμύρια τόνους πλαστικά μπαίνουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς. Αλλά η γενιά των παππούδων μου είναι μια γενιά όπου δεν υπήρχαν καθόλου πλαστικά. Οπότε, οι νέοι το καταλαβαίνουν καλύτερα, ότι τώρα 8 εκατομμύρια 8 ε, ε, ε, εκατομμύρια τόνοι μπαίνουν τόσο κάθε χρόνο στους ωκεανούς. Δηλαδή κάθε χρόνο πάει ο καθένας μας, είναι σαν να πηγαίνει ο καθένας μας κάθε μέρα στην παραλία και να πετάει τρεις πλαστικές σακούλες στη θάλασσα. Ο Μπόγιαν Σλάτ είναι αυτός που κατάφερε οι άνθρωποι να το εξετάσουν. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, κάποια στιγμή συζητούσα με τα παιδιά μου και άκουσαν ε, κάποιες συζητήσεις που κάναμε εδώ για την προστασία των δεδομένων, των προσωπικών δεδομένων των ε, πολιτών. Τα παιδιά μου δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ γι' αυτό. Μια μέρα μου είπαν, μα μπαμπά, έχουμε κάποιον YouTuber, ο οποίος μας λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να σταματήσει το ίντερνετ. Και επειδή έρχονται σε επαφή διαφορετικά με το YouTuber από ότι έρχονται σε επαφή με εμένα ε, επηρεάστηκαν από αυτά που έλεγε. Νομίζω ότι ο Μπόγιαν Σλάντ έχει διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με τους νέους. Οπότε, προσπαθούμε στον τομέα αρμοδιοτήτων μου να εξετάσουμε τη δουλειά του Μπόγιαν Σλάντ για να τη μιμηθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αν γίνεται. Δημιουργήσαμε τις αποστολές για την Ευρώπη, έτσι τις ε, ονομάσαμε και θα ήθελα μία από τις αποστολές να είναι για αντιμετώπιση των προβλημάτων των ωκεανών. Αλλά δεν θα πρέπει να είναι γενικόλογοι να πούμε ότι θα χρηματοδοτήσουμε τα θέματα των ωκεανών. Πρέπει να μιλήσουμε πολύ συγκεκριμένα στους συμπολίτε μας. Πρέπει να τους πούμε τι θα κάνουμε, πώς θα καθαρίσουμε τους ωκεανούς. Και αυτό είναι διαφορετικό τρόπος επικοινωνίας. Το είπε και ο συνάδελφός μου, ο Καρμένο. Έτσι χρειάζεται να επικοινωνήσουμε τη γενιά σας. Άρα χρειαζόμαστε τη βοήθειά σα να μας πείτε πώς να αλλάξουμε την επικοινωνιακή μας πολιτική. Και η συγκυρία είναι κρίσιμη, διότι επίκυνται οι ευρωεκλογέ. Ο κόσμος έχει αλλάξει τόσο πολύ όμως. Όταν ήρθα στις Βρυξέλλες το 2014, η κατάσταση ήταν εντελώ διαφορετική. Είχαμε τα προβλήματα των ψευδών ειδήσεων, είχαμε ορισμένους που λέγανε ότι οι ειδικοί δεν μας βοηθάνε. Ενώ τώρα η κατάσταση έχει αλλάξει. Οι πολιτικοί πρέπει να λάβουν υπόψη τη γνώμη σας, αλλά αυτό εξαρτάται από εσά. Εσείς πρέπει να πείτε στους πολιτικούς τι θέλετε, τι επιδιώκετε. Και αυτό βλέπω κάθε Παρασκευή που είμαι στο γραφείο μου να συμβαίνει. Πρέπει να καταλάβουν οι πολιτικοί ποια είναι τα σημαντικά θέματα. Ότι δεν αρκεί να λένε οι πολιτικοί ότι κάτι θα κάνουν. Πρέπει να τους πιέσετε πώς θα καθαρίσετε τους ωκεανούς, ε, πότε θα το κάνετε, με ποιες τεχνολογίες, ποιος θα τον αναλάβει. Γιατί σε τελευταία ανάλυση εξαρτώμεθα από τους ωκεανούς. Περισσότερο από όλοι πιστεύουμε. Η Σίλβια Ρέλ, την οποία αγαπώ πάρα πολύ, είπε και καταλήγω ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε θαλάσσια όντα. Δεν ζούμε μέσα στη θάλασσα, είπε, αλλά εξαρτώμεθα από τους ωκεανούς σαν να ζούσαμε μέσα στο νερό. Αυτό ακριβώς θα ήθελα να σας πω ως μήνυμα. Ότι είμαστε εδώ, μπορείτε να βασιστείτε σε μας, θα ακούσουμε τα αιτήματά σας και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε στην επόμενη περίοδο, όπως κάναμε και σε αυτή την περίοδο. Και θέλω να, να συγχαρώ τον συνάδελφο Καρμένου και το Κοινοβούλιο, την κυρία Μάισνερ, Κάναμε πολλά νομίζω. Αλλά δεν ενημερώσαμε, δεν τα παρουσιάσαμε σωστά στην κοινή γνώμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σα Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε και πραγματικά το νιώθουμε πόσο σας συναρπάζω νεοκένου. Δεν ξέρω, ίσως ε, επειδή είστε από την Πορτογαλία όπως και Επίτροπος ε, Καρμένου Μπέλα από τη Μάλτα. Ε, εγώ θέλω να αναφέρω την Ματσέλα Χάνς, γιατί αναφερθήκατε εσείς σε ένα Ολλανδό. Είναι φοιτητρία από το Άχεν, ε, μπορεί να μην την γνωρίζετε. Την ανέφερα όταν έκανα την εισαγωγή μου ομιλία. Ίσως να έχει βρει έναν τρόπο να ξεφορτωθούμε τα πλαστικά. Της αρέσει να κάνει καταδύσεις και πραγματικά όταν είδε πόσο πλαστικό υπάρχει μέσα στη θάλασσα είπε δεν μου αρέσει αυτό θέλω να το αλλάξω και έτσι δημιούργησε μια πλατφόρμα πλατφόρμα μαζί με κάποιους ε, μηχανολόγους, μηχανικούς από το Πανεπιστήμιο με την ιδέα ε, ότι τα μικροπλαστικά με τα κύματα και τα ρεύματα ε, ενώ είναι στην επιφάνεια κανονικά μπορούν να βουλιάξουν στο βυθό. οπότε αν κάπως με ένα είδος πλατφόρμας που μπορούμε να κάνουμε τα νερά να γαλινέψουν και μπορούν να ανέβουν στην επιφάνεια τα πλαστικά, θα μπορούσαμε ίσως να τα ε, περισλέξουμε πιο εύκολα. Είναι ενδιαφέρουσε ιδέε σαν αυτή του Μπόγιαν Σλάντ ή ε, αυτή τη ε, φοιτήτρα για την οποία σα ε, μίλησα εγώ. Επειδή μιλήσατε και για την κοινωνία, αυτό το θεωρώ και εγώ σημαντικό. Φυσικά και εμεί είμαστε σημαντικοί, το Κοινοβούλιο, η Κομισιόν, αλλά η κοινωνία είναι αυτή και αυτό με κάνει να ε, Σα συστήσω και την επόμενη μα ομιλήτρια, Ζενεβιέβ Πόν, από το Γραφείο των Βρυξελών του Ινστιτούτου Ζακ Ντελόρ, μια από τι ομιλήτρε που εκπροσωπεί την κοινωνία ακριβώ. Ζενεβιέβ, έχει το λόγο, παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πολύ, και Ζήνε. Ευχαριστώ και τον Καρμένου για την πολύ σημαντική αυτή πρόκληση που μου απευθύνεται να μιλήσω. Σήμερα θέλω να σας καλησπερίσω όλες και όλους, κυρίες και κύριοι, κυρίως όμω τη νέα γενιά που εκπροσωπείται τόσο καλά εδώ. Είναι προνόμιο για μένα να απευθυνθώ στην ε, συνέλευση αυτή και είναι και πάρα πολύ επίκαιρο. Η παρουσία μας εδώ είναι άκρος επίκαιρη λίγες ημέρες μετά από τη διαδήλωση ενός 1.500.000 νέων ε, που διαδήλωσαν κατά της κλιματικής αλλαγής. Ε, πρέπει να δράσουμε και εμείς. Αρκετές ε, ε, είναι οι συμφωνίες και οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει και σίγουρα αυτό θα μας κρατήσει ε, σε δουλειά για δεκαετίες ολόκληρες. Ο ωκεανός είναι η καρδιά του πλανήτη και του κλίματος. Είναι η πηγή ζωής στον πλανήτη. Ουσιαστικά μας προσφέρει την αναπνοή μας, τον αέρα που αναπνέουμε. Δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται καθημερινά στους ωκεανούς για την επιβίωσή τους. Η προστασία τον ωκεανό λοιπόν δεν είναι επιλογή, σημαίνει επιβίωση. Και αν ο ωκεανός ε, είναι υπεύθυνο για την υγεία του πλανήτη, τότε ο νότιος ωκεανός είναι η καρδιά ε, του ωκεανού. Μιλάμε για ισχυρά πολικά ρεύματα ε, γύρω από την Ανταρκτική που ουσιαστικά τροφοδοτούν τον ωκεανό με πλούσια θρεπτικά ε, συστατικά νερά. Η θαλάσσια βιοπικιλότητα μας ε, παρέχει έμπνευση, οξυγόνο, τρόφιμα. Η πηγή της είναι ο Νότιος Ωκεανός. για όσο μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου, πάντοτε με ε, τραβούσε με ήλκυε ο ωκεανός. Ε, έζησα την παιδική μου ηλικία στην Τινησία, δίπλα στη θάλασσα. Και μερικές από τις ε, πιο ε, πρώιμες μνήμε μου είναι ο καιρός που περνούσαμε με την οικογένειά μου στην Ακροθαλασσιά. Έκτοτε έκανα καταδύσεις ε, σε πολλά μέρη, σε όλο τον κόσμο και πάντοτε με κατέπλησε η ομορφιά του ωκεανού, αλλά με ανησυχούσε ταυτόχρονα βαθύτατα η υποβάθμισή του. Είτε στη χώρα μου, την πατρίδα μου, όπου οι χελώνες πεθαίνουν επειδή έχουν καταπιεί πλαστικό, ή στο κορελγενές τρίγωνο, όπου υποβαθμίζεται με πολύ γοργό ρυθμού ρυθμού ή βιοπικιλότητα. Όταν ήμουν επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Γραφείου του ΒΒΕΦ, αποφάσισα για όλου αυτού του λόγου να ενισχύσω τη δράση μα ε, για την προστασία των ωκεανών και πιο πρόσφατα, όταν ε, με είχαν προσκαλέσει να συμμετάσχω σε μια ομάδα ε, υψηλού επίπεδου άσκηση επιρροή για τη στήριξη του ε, Νότιου Ωκεανού δεν δίστασα ούτε μια στιγμή. Είμαστε η Ανταρκτική 2020, μια ομάδα ε, έξι εξαμελής από όλο τον κόσμο. Στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τον Νότιο Ωκεανό, τα νερά που ε, βρέχουν την Ανταρκτική. Είναι πάρα πολύ πλούσιο περιβάλλον αυτό του Νότιου Ωκεανού, πιγκουίνι, φάλαινες, φώκες, σε ένα οικοσύστημα που βασίζεται ε, σε πολύ μικρό αλλά πάρα πολλών ειδών κρύλ ε, βιοπλακτών ε, και χιλιάδες επιστήμονες μελετούν αυτό το κρύλ. Το 1959 στην στο αποκορύφωμα του ψυχρού πολέμου, αποφάσισαν ε, παρόλα αυτά ε, οι χώρες ε, να θεωρήσουν την Ανταρκτική ένα χώρο ειρήνης και επιστήμης. Ήταν μια πολύ γενναία πράξη και δείχνει ότι τελικά μπορούν οι πολιτικές να επηρεαστούν από την Ήπειρό μας και τα νερά της. Τα 25 μέλη της Κομισιόν για τις Επιτροπής για τη Διατήρηση των Πόρων της Ανταρκτικής έχουν δεσμευτεί ακριβώς για αυτό το σκοπό. Να προστατεύσουν δηλαδή ε, τον ε, Νότιο Ωκεανό. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος αυτής της Επιτροπής. Και όλα δείχνουν ότι η καλύτερη δυνατή προστασία του Νότιου Ωκεανού είναι με τη δημιουργία ε, προστατευμένων θαλάσσιων περιοχών μεγάλης κλίμακας. Αυτό μα ζητούν οι νέοι, να προστατεύσουμε τον Νότιο ωκεανό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προτείνει δύο σημαντικές μεγάλες προστατευόμενε περιοχές στον Νότιο ωκεανό, την Ανατολική Ανταρκτική και την θάλασσα Βέντελ. Η ε, πρόταση για την Ανατολική Ανταρκτική μιλάμε για ένα εκατομμύριο τετραγωνικά χιλιόμετρα. Πρώτα έγινε από τη Γαλλία το 2011 και περιμένουμε πολύ, ήδη έχουν περάσει χρόνια. Ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο. Πρέπει να προστατεύσουμε τώρα τον Νότιο Ωκεανό και καθυστερούμε, έχουμε προβλήματα όχι λόγω έλλειψη σπόρων, τεχνολογία ή επιστήμης, αλλά γιατί ε, την δράση αυτή την ε, επηρεάζουν ε, τα γεωπολιτικά και εθνικά συμφέροντα που θολώνουν αυτά τα παρθένα νερά. Τι περιμένουμε λοιπόν για να δράσουμε. Το 2015 ο Μπαράκ Ομπάμα έδειξε ότι ναι, είναι μεν δύσκολο να στατεύσει κανεί τον Ατοκιανό, μπορεί όμω να γίνει. Είχε μιλήσει λοιπόν ο Μπαράκ Ομπάμα ε, με τον ηγέτη της Κίνας, τον Σιζιν Jinping, και κατάφερε να υποστηρίξει η Κίνα τη δημιουργία μια θαλάσσια πρωτευόμενη προχής στη θάλασσα Ρος, στο Νότιο Ωκεανό. Και την επόμενη χρονιά, με την ρωσική αυτή τη φορά υποστήριξη, επετέχθη συνένεση για την ε, χάραξη των προσδιορισμό τη μεγαλύτερη στον κόσμο θαλάσσια πρωτευόμενη περιοχή στον πλανήτη. Πρέπει τώρα να δράσει φέτος η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γαλλία. Δεν μιλάμε για πυρηνική φυσική. Ε, ο Καρμένου Βέλα, η Φεντερίκα Μογκερίνο, ο Ντόναλτ Τούσκ έχουν δεσμευτεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προστατεύσει τον Νότιο Ωκεανό. Ο Σι ε, έρχεται στην Ευρώπη, ε, στο Μονακό αρχικά, μετά στο Παρίσι και ενδεχομένως να μεταβεί και στις Βρυξέλλες εν συνεχεία. Το σημερινό μου μήνυμα, το μήνυμα από την ομάδα Ανταρκτική 2020, το μήνυμα από τους ε, νέους που είναι εδώ παρόντες σήμερα είναι πρέπει να δράσουμε τώρα για το κλίμα και για την απώλεια της βιοπικιλότητας. Και για να το πετύχουμε πρέπει να προστατεύσουμε τον Νότιο Κιανό. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ζενεβιέβ. Νομίζω ότι όλοι θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε την Ανταρκτική μεταξύ άλλων. Τώρα ε, έχουμε και την Ντανιέλα Φερνάντες, δεν μπόρεσε όμως να μεταβεί. Έχουμε δύο άλλους εκπροσώπους, νέους, ε, Νίλε Φαν Χόιβέγγεν, που ε, είναι εκπρόσωπος ε, της ε, Ολλανδόφωνης κοινότητας του Βελγίου και ο Σεμπαστιάν Βιλμάρτ, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της γαλλόφωνης, ε, του Γαλλόφωνου Συμβουλίου Νεότητας του Βελγίου. Η Νέλε έχει το λόγο πρώτο. Σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε το λόγο. Εδώ εκπροσωπούμε τα συμβούλια του Βελγίου νεο... νεότητας και θέλουμε επίσης να θίξουμε ένα ζήτημα ύψης της σημασίας, το φυσικό περιβάλλον μας, το σπίτι μας, το μέλλον μας, την προηγούμενη εβδομάδα πάνω από ένα εκατομμύριο νέοι βγήκαν στους δρόμους έτσι ώστε να ληφθούν θαραλέα μέτρα σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές. Δεν πρόκειται για τα παιδιά μας ή για τις επερχόμενες γενναίες. Πρόκειται για μας, για το δικό μας μέλλον. Η υγεία και η ευημερία της ανθρωπότητας σχετίζεται άμεσα με το περιβάλλον μας. Η υπερθέρμανση του πλανήτη ε, έχει θερμάνει τους ωκεανούς ανά μία ατομική ε, βόμβα το δευτερόλεπτο. Δυστυχώς ε, χάνεται, πεθαίνει η θαλάσσια ζωή. Αν δεν σταματήσουμε τις εκπομπές, η Αρκτική θα είναι κατά πέντε βαθμούς ε, θερμότερη μέχρι το τέλος του αιώνα. Μιλάμε για ανεκτά επίπεδα έτσι ώστε ο πολιτισμός να επιβιώσει. Μέχρι το 2100 ο πληθυσμός θα έχει αλλοιωθεί σε σχέση με σήμερα. Σκεφτείτε ποια θα είναι μία εικόνα δορυφόρου του μπλε πλανήτη που δεν θα είναι πλέον μπλε. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε τις ε, κοραλιογενείς ε, εκτάσεις που αποτελούν ένα 25% της θαλάσσιας ζωής. Όμως το IPCC δείχνει ότι με αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 βαθμό θα, χαθούν, θα χαθεί ένα πολύ υψηλό επίπεδο κοραλιογενής ευλάστησης. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα ορυκτά καύσιμα χρησιμοποιούνται κατά πολύ στις χώρες του ΩΣΑ Κάτι το οποίο ε, δείχνει ότι το δικαίωμα στο ε, νερό πρέπει να υπάρχει, καθώς και να απαγορευτεί η γλυφοσάτη. Πώς ε, δεν μπορείτε να είσαστε δραστήριοι. Η Ευρώπη έχει αναλάβει πρωτοβουλίες, αλλά αυτό δεν θα μας περισσώσει. Μιλάτε για την γαλάζια οικονομία. Αυτός ο νέος όρος είναι μία, δεν θα είναι δεν θα πρέπει να είναι μία σήμανση, θα πρέπει να μας οδηγήσει σε συγκεκριμένες πρακτικές που σχετίζονται με τους ωκεανούς. Δεν θα πρέπει να προωθήσουμε δράσεις που είναι επιζήμιες στο περιβάλλον. Θέλουμε να δεσμευτείτε όλοι προς αυτό. Οι ωκεανοί είναι ένα νέο ελντοράντο, είναι πόροι, είναι αναψυχή είναι ε, θρεπτικά συστατικά μεταξύ πολλών άλλων, από τα οποία εξαρτώμαστε πλήρως και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Η προστασία των ε, οικοσυστημάτων των ωκεανών είναι ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές για την επιβίωση βιώσιμων οικοσυστημάτων για τους ανθρώπους, τη φύση και τις επιχειρήσεις. Σας παρακαλούμε να το κάνετε σοβαρά, σας προτρέπουμε να ισχύσουν οι κανόνες αλίας στον τομέα αλίας για να μην γίνεται χρήση πλαστικών στις ε, προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. η παγκόσμια διακυβέρνηση των ε, ωκεανών δεν θα αρκέσει από μόνη της. Η καταπολέμηση Σημαντική αλλαγή. η καταπολέμηση της φτώχειας ε, είναι μια παγκόσμια πρόκληση. Πρέπει να υπάρξει διαρθρωτική δράση. Πρέπει να επαναδιαμορφωθεί το σύστημα ανάλογα με την φυσική, φυσιολογική πραγματικότητα με την φυσική πραγματικότητα του πλανήτη και των συμπολιτών. Το θέμα δεν είναι να καθαρίσουμε μόνο του ωκεανού. Είναι να σταματήσουμε να του μολύνουμε. Ξέρουμε την κατάσταση. Ξέρουμε και τις λύσεις. Αλλά ε, τα παραβλέπετε όλα αυτά. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας υπενθυμίσω κάποια θέματα. Ε, πρέπει να μιλήσουμε για τη χρηματοδότηση. Θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε το θέμα της φορολογικής δικαιοσύνης όχι μόνο με λόγια αλλά και με έργα. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φόρο για τον άνθρακα. Θα πρέπει η Κομισιόν ε, να καταπολεμήσει επίσης την ε, φόρο αποφυγή κατά προτεραιότητα στην επόμενη θητεία και να θέσει ένα τέρμα στο φορολογικό ντάμπινγκ και τα κοινωνικά ζητήματα βέβαια είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να είναι γνώμονας στις ε, εν λόγω πρωτοβουλίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη πρέπει να υιοθετήσουν μια διαφορετική θεώρηση για τα δημοσιοοικονομικά. Η χρηματοδότηση ε, να κρίνεται με βάση το πόσο συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή να επενδύουμε εκεί που μετράει. Δεν μιλάμε όμως μόνο για επιχορηγήσεις δημοσιοοικονομικά. Πρέπει να κατανοήσουμε το εμπόριο ε, ως ένα παράγοντα που μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Δεν θα πρέπει να έχουμε δυσανάλογη συγκέντρωση πλούτου ούτε διαιώνιση ανθιγυνών τρόπων ζωής. Για παράδειγμα, μπορούμε να υιοθετήσουμε τον δίκτυο ανθρώπινη ανάπτυξη, που είναι ένα βασικό δείκτη επιτυχία και όχι απλά η ανάπτυξη με βάση το ΑΕΠ να είναι το κριτήριο. Πρέπει επίση το πολυμερέ εμπορικό σύστημα να μεταρρυθμιστεί στο πλαίσιο αυτό και οι κανόνες του ΠΟΕ, ώστε να λάβουν μεγαλύτερη προτεραιότητα περιβαλλοντικά ζητήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει κάποια μικρά βήματα προηγουμένως, όπως η πρόταση για αύξηση του ενωσιακού προπολογισμού και των ταπανών για ε, το κλίμα κατά 25%, όμως αυτό δεν αρκεί. Είναι σαφές. διότι θα πρέπει να μετριαστεί η αλλαγή του κλίματος. Θα πρέπει να δοθούν πόροι για την οικολογική μετάβαση. Για εβδομάδες κατεβαίνει ο κόσμος ε, και διαδηλώνει. Άρα χρειάζεται συστημική αλλαγή, όχι κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν αιτήματα που σχετίζονται συγκεκριμένα με του ωκεανού. Ζητούμε όμω πέραν αυτού τη διαγενειακή δικαιοσύνη και την ισότητα να την θεωρήσετε σημαντική κατευθυντήρια γραμμή για τι πολιτικέ σα όλα τα επίπεδα. Οι επιστημονικέ ε, μαρτυρίε, τεχνικέ λύσει, ε, η κρίσιμη μάζα ε, είναι κάτι που το έχουμε. Το έχουμε επιτύχει. Αυτό που απαιτείται τώρα είναι να επιδειχθεί πολιτικό σθένος και είναι η τέλεια στιγμή χρονική να γίνει αυτό, διότι η κοινή γνώμη είναι ιδιαίτερα υποστηρικτική. Το μέλλον μας είναι αυτό το οποίο παίζεται στην κυριολεξία. Έχετε λοιπόν την ευκαιρία να ε, διαλέξετε το μέρος της ιστορίας στο οποίο θέλετε να είστε. Μπορούμε να εργαστούμε μαζί για να προστατεύσουμε το μέλλον ε, και των ε, νυν και των μελλοντικών γενιών. Ας είστε κι εσείς μέλος κομμάτι Ευχαριστώ. Νέλε και Σεμπαστιά, ακούσαμε αυτά που μας είπατε, μας συγκίνησαν ιδιαίτερα και εν γέννη η συνεισφορά σας. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε Βέβαια, είναι πολύ δύσκολο να μετατρέψουμε την πολιτική σε πραγματικότητα, αλλά προσπαθούμε. Λίγη λοιπόν τώρα η, εναρκτήρια, ε, η έναρξη της διάσκεψης. Θα πάμε για την οικογενειακή φωτογραφία έξω στο άτριουμ. Πριν όμως από την οικογενειακή φωτογραφία θα έχετε ένα νέο ε, πάνελ υπό τον ε, Αλέν Καντέκ. Δυστυχώς όμως άργησε η πτήση του και γι' αυτό η Ντάρια Μάτο θα αναλάβει το επόμενο πάνελ και θα ήθελα όλοι οι πάνελιστ στη συνέχεια να έρθουν να μας αντικαταστήσουν. Άρα τώρα θα πάμε για την οικογενειακή φωτογραφία και μερικοί θα επανέλθουν. Ο Ντάριο Μάτο θα είναι ο Γκάμπριελ Μάτο θα αναλάβει το πρώτο πάνελ το οποίο θα αρχίσει σε 10 περίπου λεπτά.